Δημοκρατία και από τις 23 Ιουνίου 2010 θα λογίζεται με τους μη εγγεγραμμένους. Επίσης οι αρμόδιες αρχές ε, της Ολλανδίας με πληροφόρησαν πως ο Λουίς Μπόντες αντικαταστάθηκε από τον Λούκας Χάρτονγκ και η κυρία Ζανίν Χενής από τον κύριο Γιάν Μιλντερ από τις 22 Ιουνίου 2010. δύο από χτες. Καλώς ορίζω τους ε, νέους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού μέχρι να υπαλληθευτούν ε, οι εντολές τους ο κύριος Λούκας Χαρτόν και Γιάν Μίλντερ θα συμμετέχουν έχοντας επίσης δηλώσει πως δεν έχουν κάποια, κάποιο άλλο αξίωμα που είναι ασυμβίβαστο με αυτό του Ευρωβουλευτή. γραμματεία των μη εγγεγραμμένων